Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ όλους. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ και μία κατά. Okay. Let's start. Ξεκινάμε με το σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ισχύα. Όσοι δεν θέλουν να παραμένουν, μπορείτε να αποχωρήσετε. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως και ο αναφέρον μας παρακολουθεί μέσω διαδικτύου. Έχουμε λοιπόν την αναφορά 38-2019 από Ρουμάνο Υπήκο για τη διάκριση από πλευράς του eBay ε, για άτομα που κάνουν αγοράς μέσω Ρουμανίας. Ο αναφέρον παρακολουθεί μέσω διαδικτύου την ε, ε, Επιτροπή μας. Να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, στην κυρία Τζασμίν Μπατίστα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται λοιπόν για μια αναφορά η οποία αφορά διάκριση του eBay κατά αγοραστών από, το eBay, ε, από τη Ρουμανία, σύμφωνα με την καταγγελία του αναφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει σχετικές πληροφορίες και απάντησε ότι όντως ε, κατά την άποψή μας δεν υπάρχει άμεση παραβίαση σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση παράδοσης ε, για τους εμπόρους ε, βάσει του κανονισμού ε, για το γεωγραφικό αποκλεισμό προς το παρόν. Επομένως, είχαμε προτείνει στον αναφέροντα να το συζητήσει με τις αρχές καταναλωτή για να δει και τι ισχύει όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και τα σχετικά στοιχεία. Αυτό το οποίο συνέβη το μεταξύ και έχει και ενδιαφέρον να γνωρίζετε είναι ότι όπως ξέρετε μας επιβάλλεται υποχρέωση να παρακολουθούμε την εφαρμογή του κανονισμού και να υποβάλουμε και έκθεση. Η προθεσμία είναι στα τέλη Μαρτίου, επομένως ε, εμείς προσπαθούμε να τηρήσουμε και τη σχετική προθεσμία και έχουμε μια έκθεση και το έγγραφο εργασίας εξηγεί πώς έχει προχωρήσει ο κανονισμός μέχρι τώρα τι εμπειρία έχουμε με τον κανονισμό από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται στις 3 Δεκεμβρίου του 2018 και εξετάζουμε και ε, το ενδεχόμενο αλλαγής του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό το οποίο έπρεπε να εξετάσουμε πρωτίστως ε, είναι εάν ο κανονισμός πρέπει να επεκτηθεί και σε οπτικοακουστικά και σε άλλους ε, τομείς οι οποίοι προς το παρόν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Συγγνώμη επιλογή της παράδοσης αγαθών δεν ήταν μεταξύ αυτών που έπρεπε να εξετάσουμε καταρχήν, αλλά υπάρχουν ε, και δυνατότητες ε, αναθεώρησης του κανονισμού για το γεωγραφικό αποκλεισμό και ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την υποχρέωση. Προ το παρόν θεωρούμε ότι είναι αρκετά σαφέ ότι ο κανονισμός για το γεωγραφικό αποκλεισμό αυτός καθ' αυτό δεν ε, υποχρεώνει τον έμπορο να παραδίδει αγαθά σε κάποιες χώρες και επομένως επειδή είναι δική του επιλογή, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον έμπορο να στέλνει αγαθά στη Ρουμανία δεν έχουμε συζητήσει και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση μετά από αυτή την ανταλλαγή και δεν ε, λάβαμε και πληροφορίες για τα κατά πόσον ο αναφέρον συζήτησε με τις εθνικές αρμόδιες αρχές είναι αυτέ οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του κανονισμού. Επομένω, αν υπάρξει παραβίαση, θα πρέπει να ε, υπάρξει διαδικασία επιπαραβάση από αυτούς και η νομοθεσία φυσικά εφαρμόζεται. Εν τω μεταξύ, η Ρουμανία ενέκρινε και τη σχετική νομοθεσία, καθυστέρησαν λίγο, αλλά μόλις λάβαμε πληροφορίε ότι έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Επομένως, οι πιέσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού δεν χρειάζεται να συνεχιστούν, διότι λογικά υπάρχει πλέον ο νόμος και υπάρχει αρμόδια αρχή η οποία μπορεί να αποφασίσει επί του ζητήματος. Ε, ίσως ε, κάτι επιπλέον που θα μπορούσα να πω είναι ότι στο νέο κανονισμό CPC, ο οποίος ισχύει πλέον τώρα σε σχέση με το παρελθόν, υπάρχουν και κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία βοηθούν τους καταναλωτές ε, όσον αφορά το γεωγραφικό αποκλεισμό και σχετικές πρακτικές αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βοηθήσει ε, τον αναφέροντα και για την περίπτωση παράδοσης αγαθών ε, στη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννη. Ναι, ε, χαίρομαι που υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Για μένα ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Στο, στο εμπόριο με το ίντερνετ κάποια προϊόντα εκ των πραγμάτων ε, αποκλείοντο και έγινε η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ψηφιακός ε, κόσμος στον νούμερικό και αντιστρόφως αν αγοράσει κανείς στην ένα αυτοκίνητο στη Φιλανδία, αυτό μπορεί να, και μένω στον αρκτικό κύκλο, αυτό μπορεί να επιτρέπεται. Αλλά το θέμα είναι πώς θα πάρω το αυτοκίνητο είτε θα πάνω το πάρω ο ίδιος, είτε θα πρέπει να καλυφθούν τα κόστα μεταφοράς. Αυτό δεν έχει να κάνει με διακρίσεις. Όταν κάποιος λέει ε, ότι θα πρέπει να πάει να παραλάβει ο αγοραστής ε, ο ίδιος το αυτοκίνητό του, γιατί έτσι γινόταν στο παρελθόν. Και, με το, και ε, γι' αυτό το λόγο ορισμένα προϊόντα έπρεπε να αποκλειθούν. Άρα το πρόβλημα εδώ είναι το θέμα της ε, πρόσβασης στο προϊόν το οποίο έχει αγοραστεί. Ίσως ε, ε, θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε ανοιχτό το θέμα για λίγες εβδομάδες και η Επιτροπή στη συνέχεια να δώσει μία απάντηση στον Τούντα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα, δεν πρόκειται για διακρίσεις εδώ. Όπως είπε η Επιτροπή, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις για την, τις online πωλήσει. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη δουλειά, όντως. Ο αναφέρον ε, έχει υπογραμμίσει την εμπλοκή των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες και το ζητά την, τονίζει ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί, πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, επαναξετάζοντας τον κανονισμό, για να δούμε κατά πόσον μια νέα προσέγγιση θα δώσει περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές και τους πολίτες. Προτείνω να μείνει ανοιχτή, λοιπόν, η διαδικασία. Στα ρουμανικά πρόεδρε θα μιλήσω. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το οποίο έχει θέσει ο αναφέρον. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν πρόκειται μόνο για αγορές eBay εδώ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγορές online Ορισμένες φορές ε, όντως επιφέρουν κάποιες διακρίσεις ε, σε πολίτες ε, από χώρες μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να εξτάσουμε περισσότερο τα θέματα αυτό και με ένα πιο διαρθρωμένο τρόπο, γιατί δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνεί ότι ορισμένες χώρες μέλη υφίστανται κάποιες ε, διακρίσεις όταν ε, μιλούμε βεβαίως για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Και εφόσον ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να προσπαθήσει να κάνει περισσότερα πράγματα προκειμένου να αποφευθούν τέτοιες διακρίσεις. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι πολλοί πολίτες Ε, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ε, πάσης ε, φύσεως ξένα μέσα πληρωμής γιατί η ρουμανική πιστοτική κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές σε τέτοιες πλατφόρμες αγοράς προϊόντων online. Και βεβαίως υποστηρίζω την ε, πρόταση του συναδέλφου το θέμα αυτό να παραμείνει ανοιχτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Αφού ακούσαμε την Επιτροπή και τα μέλη, η πρότασή μας είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να περιμένουμε την Επιτροπή να τελειώσει τη μελέτη της. Μας είπε ότι θα τελειώσει τον Μάρτιο. Επόμενο σημείο. 1100 67-2018 από έναν Έλληνα πολίτη για την εμπορία προϊόντων Huawei στην Ελλάδα και την Ένωση και την αναθεωρήση όλου του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στην Ένωση για να προσφέρουν ασφάλεια και να καταργήσει, να εμποδίσει κατασκοπευτικά δίκτυα. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Ο κ. Φεράρα θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που δίνετε στην Επιτροπή την ευκαιρία να μιλήσει εκτενέστερα για την απάντηση αυτή, δίνοντας μια ενημέρωση για την διαδικασία μετά την υποβολή των παρατηρήσεων της Επιτροπής. Καταρχά να τονίσω ότι εμείς θέλουμε πάντα να προωθήσουμε ένα ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και εμπορευόμενους να υποφεληθούν ελεύθερα των δικαιωμάτων που παρέχει η ενιαία αγορά. Παρακολουθούμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μόνιμα για να βλέπουμε κατά πόσον η επιχείρηση αυτή συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζουμε ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με, τον, με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα για την ασφάλεια των του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, ανάπτυξη του 5G, της ε, σύνδεσης επόμενης γενιάς στα κράτη-μέλη. Και αποφάσισε να εκδώσει μια σύσταση, ε, στις 26 Μαρτίου έγινε αυτό, που θέτει ακριβώς ένα πλαίσιο διαδικασιών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτίμηση των μέτρων ε, προστασίας από παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα. Μετά από αυτή τη σύσταση, τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με, με την Επιτροπή και την ΕΝΙΖΑ έχουν ξεκινήσει μία δράση για να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της επιτόπου. Τα κράτη-μέλη επίσης ε, εξέφασαν το ενδιαφέρον να, επι... να λειτουργήσουν ως πρωτοπόροι στην εφαρμογή της σύστασης με μια σειρά σημαντικών μέτρων. Τα κράτη-μέλη μέσω της σύστασης έπρεπε να υποβάλουν, για παράδειγμα, ένα, μια εθνική αξιολόγηση κινδύνου μέχρι το καλοκαίρι πέρσι. Με χαρά είδαμε ότι όλα τα κράτη-μέλη το έκαναν. Βάση αυτής της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου στις 9 Οκτωβρίου τα κράτη-μέλη που ήταν ε, μέλη της ομάδας εργασίας NIS παράλληλα με την ΕΝΙΣΑ και την Κομισιόν δημοσίευσαν ένα συντονισμέ... μια συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο ένωσης. Αυτή η αξιολόγηση κινδύνου εξέτασε ποιες είναι οι τάσεις, ποια είναι τα τεχνικά και μη τεχνικά τα σημεία στα δίκτυα 5G και παρουσίασε μια σειρά 5 σεναρίων κινδύνου. Τα ευρήματα είναι ότι οι κύριες προκλήσεις των δικτύων 5G οφείλονται κατά βάση στις ε, ιδιαίτερα καινοτόμες τεχνολογίες, κυρίως αυτές που βασίζονται σε λογι... σε... στον εξοπλισμό λογισμικού. Καινοτομία δηλαδή σε σχέση με παλαιότερα δίκτυα 4G και τον βασικό, σημαντικότερο ρόλο των προμηθευτών στην διαμόρφωση και η κατασκευή των δικτύων 5G, 5G. Αυτό ήταν ένα βασικό ορόσημο. Το επόμενο ορόσημο που τα κράτη-μέλη ή η Επιτροπή και ενίσα εξετάζουν είναι η επιτροπη και εξεταζουν ενός μιας εργαλειοθήκης μέτρων περιστολής του κινδύνου, μετριασμού του κινδύνου. Θα ετοιμαστεί σύντομα. Μία ένα από τα βασικά μέτρα της Επιτροπής έχει να κάνει με την πιστοποίηση. Έχουμε ένα εργαλείο τώρα που ε, διαμορφώνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας με βάση και την νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια στην Ένωση που υιοθετήθηκε πέρσι τον Ιούνιο. Θα δούμε τώρα μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πιστοποίηση ως ένα μέτρο μετριασμού του κινδύνου. Παράλληλα με άλλα πιθανά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη της Επιτροπής τώρα. Ποιος θέλει να παρέμβει. Ο κύριος Αλίμπα. Εγώ συμφωνώ πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μια επιχείρηση πρέπει να ενταχθεί νομίμως στην εσωτερική αγορά, υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τους καταναλωτές μας, ιδιαίτερα όταν ελοχεύει ο κίνδυνος ε, για την προστασία των δεδομένων τους και την ε, ασφάλεια. Καταρχάς ε, θα ήθελα η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και επίσης ταυτόχρονα να ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει και μια συνέχεια για το πώς ε, τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν το θέμα της ε, των παρόχων από τρίτε χώρες για τα δίκτυα 5G και επίσης να το στείλουμε και στην Επιτροπή ΕΜΚΟ για γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, κύριος Βίνθε. Ευχαριστώ το κυρία Πρόεδρε και ε, εξ ονόματος του ΕΛΚ και εμείς ε, θα θέλαμε να προτείνουμε να κλείσει αυτή η αναφορά. Δεχόμαστε την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύουμε ότι η πρόσβαση της ε, Huawei στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εξοπλισμό ανάπτυξης τεχνολογίας 5G είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα Ξεκίνησε από τις Ηνωμένε Πολιτείες το όλο ζήτημα και στη συνέχεια όλοι ε, στις Πολιτείες εξετάζουν τα θέματα αυτά, αλλά όσον αφορά την αναφορά, ήδη βρισκόμαστε πολλά βήματα μπροστά και θεωρώ ότι μπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση, διότι έχουμε εξασφαλίσει και μια σωστή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Προεδρία πάντα προσπαθεί μετά από τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν έχουμε παρουσία του αναφέροντος και επίσης ε, ακούσαμε και τα όσα είπαν τα μέλη της Επιτροπής. Προσπαθώ πάντα λοιπόν να ε, δίνω μια ισορροπημένη λύση. Και επειδή το ΕΛΚ ζήτησε να κλείσουμε το θέμα και οι σοσιαλιστές ζήτησαν να παραμείνει ανοιχτό και δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να θέλει το λόγο ούτε από κάποια άλλη πολιτική ομάδα, η πρόταση της Επιτροπής μας είναι να θεωρήσουμε ότι έκλεισε η αναφορά, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ή άλλως ε, προωθεί την ε, ισότιμη μεταχείριση για όλους τους παρόχους εξοπλισμού 5G και φυσικά εξασφαλίζουν και ότι θα υπάρχει παρακολούθηση του σχετικού δικτύου. Κλείνουμε λοιπόν, προτείνουμε να κλείσει γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί και εργάζεται για να προστατεύσει την κυβερνοασφάλεια και ε, να υπάρχει και ε, ισότιμη μεταχείριση σε όσου δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συμφωνείτε λοιπόν θα κλείσουμε την αναφορά. Περνάμε στο σημείο 20 που είναι η αναφορά 1151-2018 από τον Χόλκερ Βάγνερ, Γερμανό πολίτη, για μια ανεξάρτητη επιστημονική έκθεση για τους καταγεγραμμένους κινδύνους για την υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ε, έτοιμα για αναβολή της εφαρμογής του ε, δικτύου 5G να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, ε, γιατί δεν είναι εδώ αναφέρον. Ο κύριος Φρανς Κάρχερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνοψίσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι το άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, δεν δίνει εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει νομικά δεσμευτικά μέτρα για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για λόγους ε, δημόσιας υγείας. Παρά το γεγονό ότι είναι περιορισμένη η αρμοδιότητά μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κάποια όρια στο Συμβούλιο το 1999 και το ε, Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση 1999-519 αλλά φυσικά η σύσταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Έχουμε όμως και ε, δύο εκθέσεις εφαρμογής και από αυτές τις εκθέσεις εφαρμογής ε, μαθαίνουμε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά όρια και κάποια κράτη-μέλη έχουν ακόμα και πολύ πιο χαμηλά όρια, μέχρι και 10 φορές πιο χαμηλά από αυτά τα οποία προβλέπονται από τη σύσταση. Η σύσταση βασίζεται στις κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, της ε, Διεθνούς Επιτροπής για τη μειονίζουσα προστασία, μάλλον της μειονίζουσας ακτινοβολίας και αυτή τη στιγμή γίνεται μια αναθεώρηση, η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση έγινε το 2018 και εξ όσων γνωρίζουμε οι νέες αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ε, σταλεί σε επιστημονικό περιοδικό και είναι σε διαδικασία αναθεώρησης, επομένως θα δημοσιευθούν ε, προσεχώς. Μόλις ε, είναι διαθέσιμες δημοσίως αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Η μία περίπτωση με τη βοήθεια της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία, για περιβαλλοντικούς και αναδυόμενους κινδύνους που ε, είναι μια επιτροπή με την οποία διαβολευθήκαμε στο παρελθόν και υπάρχει και η δυνατότητα να ε, διαβουλευτούμε το μηχανισμό επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει περισσότερο αλλά είναι ένα δίκτυο 150 ακαδημιών και ε, ιδρυμάτων ανά τον κόσμο και περιμένουμε και ασφαλείς επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από αυτούς. Τώρα, η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ε, γνωμοδοτεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά, μας έχει δώσει διάφορες γνωμοδοτήσεις, η πιο πρόσφατη το 2015, και υπάρχουν τρία βασικά συμπεράσματα, τα οποία θα ήθελα να σας συνοψίσω εδώ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα όρια τα οποία συστήνονται από το Συμβούλιο εξακολουθούν να ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη Ένα όμως από τα συμπεράσματα ήταν ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για σταθμισμένη έρευνα, διότι ορισμένες φορές δεν είναι επαρκής η ποιότητα της ε, έρευνας. Στην αναφορά αυτή υπήρχε και μια κάποιες μορφής κατηγορία ότι το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής δεν είναι αμερόληπτο και ότι η επιστημονική βιβλιογραφία επελέγει σκοπίμως ε, για τη συγκεκριμένη σύσταση. Εδώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων για οποιοδήποτε μέλο της Επιτροπής ή της ομάδας εργασίας του και επίσης ε, έχει υπάρξει ήδη μια περίπτωση ε, για ισχυρισμούς για έλλειψη αμοροληψίας, ε, η οποία παραπέμφθηκε και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και ο Διαμεσολαβητής μετά από εξέταση του θέματος ε, θεώρησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε καλές διοικητικές πρακτικές σε αυτές τις περίπτωση. Θα ήθελα επίσης να συνοψίσω και κάποια επιχειρήματα όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Καταρχάς, οι κατευθυντήριες γραμμές και η σύσταση του Συμβουλίου εφαρμόζουν ήδη την αρχή της ε, πρόληψης, διότι υπάρχουν παράγοντες ασφαλείας, ε, οι οποίοι είναι μέχρι 10 φορές για τους εργαζομένους και 50 φορές για το ευρύ κοινό, που σημαίνει ότι τα όρια έκθεσης, τα οποία καθορίζονται στη σύσταση, είναι μέχρι και 50 φορές ε, χαμηλότερα από τα επίπεδα τα οποία βάσει επιστημονικών γνώσεων αρχίζουν να υπάρχουν ε, αποτελέσματα σε ανθρώπινους ιστούς. Επίσης, η νέα τεχνολογία 5G ε, χρησιμοποιεί αντίστοιχες ε, συχνότητες με το 4G. Επομένως, η χρήση της ίδιας συχνότητας καλύπτεται και αυτή από τη σύσταση και από τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα νέα ε, έξυπνα κινητά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ε, ε τεχνολογία 5G σημαίνει ότι έχουν κάποιες δυνατότητες εντός του τηλεφώνου που σημαίνει ότι έχουμε εκπομπή ισχύους μόνο ε, σε περίπτωση επικοινωνίας μεταξύ για παράδειγμα κινητών τηλεφώνων και μιας μικρής κεραίας Δεν είναι συνεχής η εκπομπή της ακτινοβολίας. Από κάποια ε, δυνατότητες που έγιναν στην Αυστραλία, ε, είχαμε εκπομπή στη μέγιστη ισχύ και τα άτομα τα οποία συμμετείχαν εξετέθηκαν σε λιγότερο από 1% από τα όρια τα οποία έχουμε καθορίσει στη σύσταση. Και επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν την ίδια τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, γιατί είναι η βασική στόχη ε, τα, τα βασικά εργαλεία έκθεσης ε, χρησιμοποιώντας ακουστικά ε, και να σε αυτή την περίπτωση έχουμε λιγότερη ισχύ και λιγότερη έκθεση. Και επίσης θα πρέπει να φέρουμε και στην εξίσωση και τα ωφέλη τα οποία περιμένουμε από την εφαρμογή των δικτύων 5G και της σχετικής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, όσον αφορά ιατροτεχνολογικές συσκευές και τεχνητή νοημοσύνη. Ε, συνοψίζοντας λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι αμερόληπτο, υπάρχουν αυστηροί κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται και οι ισχυρισμοί αυτοί είναι βάσιμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό που ζητάει άλλωστε είναι που ζητάει ο αναφέρον, θα χρησιμοποιήσει τις επιστημονικές γνώσεις για να κάνει μια εις βάθος ανάλυση και αναθεώρηση για τη σύσταση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γκρικά. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί στο μέτρο που εξελίσσεται η τεχνολογία θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεχής ε, αναθεώρηση και εξέταση η οποία αναλαμβάνει υπόψη της τόσο το περιβάλλον και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Προφανώς ο σκοπός αυτής της αναφοράς δεν είναι να τεθεί αναμφιβόλο η χρησιμότητα της ε, τεχνολογίας 5G, αλλά σκοπός της αναφοράς είναι απλώς να βάλει στο τραπέζι περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την απάντησή του και θα πρέπει να δούμε ότι η Επιτροπή έχει βασιστεί στα επιστημονικά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί τα δίκτυα 5G. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις ε, επιπτώσεις που έχουν τα δίκτυα αυτά στην ανθρώπινη υγεία. Τώρα ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση προπαρασκευής και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία αυτή θα έχει εφαρμοστεί τότε ε, θα πρέπει ακριβώς να εκπονηθούν οι μελέτες. Άρα λοιπόν συμφωνώ με τον αναφέροντα γιατί θα πρέπει να αναλυθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Αλλά ακόμα ε, βρισκόμαστε μέσω μιας μακράς διαδικασίας. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, οι αναλύσεις Ε, αυτά αυτές θα πρέπει να είναι πιο λεπτομεριακές. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή είναι να αφήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σαλίβα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την ε, εμπεριστατωμένη ανάλυση και παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα αυτό όσον αφορά την ε, δημόσια υγεία, θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Και παρόλο που η Επιτροπή είπε ότι υπάρχει ένα θέμα μεροληψίας ε, και βεβαίως ε, το ζήτημα αυτό έχει επικυρωθεί και από τον ε, διαμεσολαβητή. Και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε ότι η ποιότητα της έρευνας όσον αφορά τις επιπτώσεις των δικτύων 5G δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η αναφορά αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και επίση θα πρέπει να αποσταλεί στην, να παραμευθεί στην Επιτροπή ΕΜΒΗ για γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την άποψη ότι ότι εδώ θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Γιατί η Επιτροπή Προστασία από τη μη ακτινοβολία δεν είναι διεθνή επιτροπή η οποία να είναι ανεξάρτητη. Πρόκειται για μια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό οργανισμό λόμπι ε, της βιομηχανίας που δεν είναι καθόλου ανεξάρτητος. Ε, εγώ ε, θα ε, δημοσιεύσω ένα κείμενο το οποίο θα καταδεικνύει το ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων των χωρών μελών. Ε, όσον αφορά την γνωμοδότηση της ΣΥΡ, της Επιστημονικής Επιτροπής για Υγεία Περιβάλλον και Αναδιόμενους Κινδύνους, δημοσιεύθηκε το 2015 και εγώ ίδιος μελέτησα αυτή την έκθεση την αναφορά και διαπίστωσα ότι πολλές σημαντικές εργασίες οι οποίες έχουν αποδείξει τις ε, ζημίες, τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία έχουν ε, παραμεληθεί. Ε, για παράδειγμα, οι βλάβες στο DNA. Γνωρίζουμε από επιστημονικά πειράματα ότι υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι για τα ε, μαλακά κύτταρα. Και η έκθεση αυτή ανεμειγνύει τα πάντα και βεβαίως στην περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να εντοπιστούν με κίνδυνοι σε ορισμένους, σε άλλους πάλι όχι. Και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση είναι εντελώ αόριστα και σαφής, άρα δεν μας ενδιαφέρει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το συμπέρασμα, αλλά πραγματικά κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Και στην τελευταία παράγραφο της έκθεσης, μάλλον της απάντησης της Επιτροπής, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν ισχύει ότι μειώνεται η ακτινοβολία για τα συστήματα 5G στα, στις ΗΠΑ ε, έχει ανέβει το όριο. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιείται για τα 5G ε, χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια. Παρ' όλα αυτά ε, δεν μειώνεται η ακτινοβολία. Όσον αφορά τι συχνότητες θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις εδώ. Ε, στα 5G έχουμε μια, ένα μείγμα διαφόρων συχνοτήτων και δεν θα επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειε, αλλά είναι ξεκάθαρο το εξή. Η Επιτροπή Προστασία αποτιμεί η ιονίζουσα ακτινοβουλία ε, ένα εντελώς ε, δογματικό συμπέρασμα ε, ότι μόνο η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι επιζήμια. Ε, κάτι το οποίο έχει αμφισβητηθεί από πάρα πολλές, από πληθώρα επιστημονικών εργασιών. Γνωρίζουμε την, ε, τις βλάβες προκαλούνται από τις τωρινές ε, οριακές τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. σε μια Αμερικάνικη πολιτεία έγινε μια μελέτη η οποία αποδεικνύει σε αρσενικά ποντίκια την, ε, τις, ε, ζημίες, τις βλάβες που προκαλούνται από αυτά τα επίπεδα ακτινοβολίας. Και αντίστοιχε έρευνε, έγιναν και στην ε, Ιταλία και απέδειξαν, κατέληξαν τα ίδια αποτελέσματα. και στον άνθρωπο ισχύει το ίδιο οι ισχύουσες ακτινοβολίες, οι ισχύουσες σωριακές τιμές είναι ήδη ε, ζήμιες, ε, επιζήμιες και ε, κακινογόνες. Άρα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Να παρέμβω ως πρόεδρος της Επιτροπής με δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Πρώτον, Υπάρχουν, το είπε πολύ καλά ο κύριος Βίντσε από το ΕΛΚΑ. Εδώ συζητούμε νέες τεχνολογίες, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εξετάζοντας διεξοδικά τις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία των νέων αυτών τεχνολογιών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Υπάρχουν σαφή αποτελέσματα ως προς το κατά πόσον η έκθεση στα 5G δεν επηρεάζει ευάλωτες ομάδες. Δεύτερη ερώτηση. Η Επιτροπή για να, μην, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε χωρίς αμφιβολίες. Η Επιτροπή είναι σαφές ότι οι συστάσεις ε, του Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτικές για τα κρατημέλη. Μπορεί η Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση όταν, ε, ε όταν εμφανιστούν οι νέες οδηγίες από το ICNIRP. Δηλαδή, η έκθεση του ICNIRP ε, θα οδηγήσει την Κομισιόν στο να πάρει κάποια άλλη απόφαση. Ευχαριστώ. Για το πρώτο. Είναι εξαιρετικά επιστημονικό θέμα, οι σύμβουλοι μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέχρι τώρα βάσει επιστημονικών στοιχείων, όπως έχουν τεθεί, γι' αυτό δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού, ομάδες κινδύνου, επηρεάζονται αρνητικά από τις τεχνολογίες αυτές ενώσω τα όρια που, θέτουν, που θέτει η σύσταση τηρούνται. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχουμε, έχουμε πολύ περιορισμένα στοιχεία για τη νέα αυτή τεχνολογία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επιδημιολογικά θα γίνει αυτό, διότι η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται ακόμα. Για το δεύτερο σημείο, σε λίγες εβδομάδες μόνο θα βγει η νέα αυτή δημοσίευση. Έχει ήδη σταλεί στην επιστημονική κοινότητα και στο περιοδικό Health and Physics από πέρσι και περιμένουμε να δημοσιευθεί ο Σονούπο. Θα εξετάσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Είτε την επιστημονική κοινότητα είτε τον μηχανισμό επιστημονικής συμβουλής. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Αν δεν κατάλαβα καλά, αν κατάλαβα είπατε ότι δεν χρησιμοποιείται η παράμε... ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν στοιχεία βλάβης γιατί δεν χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Όταν αναπτυχθεί πλήρως το δίκτυο αυτό, τότε θα δούμε αν υπάρχουν επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα δεν γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης για τις ευάλωτες ομάδες, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως το δίκτυο και η Επιτροπή περιμένει την έκθεση του ICNIRP για να συνεχίσει την μελέτη για τον αντίκτυπο στην υγεία όταν η νέα αυτή τεχνολογία αναπτυχθεί πλήρως. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι τεχνικό ζήτημα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Μου ζήτησαν να αφήσουμε ανοιχτή τη διαδικασία, αλλά δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να μόνο να αφήσουμε ανοιχτή τη διαδικασία. Πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα. Είμαι δικηγόρος εγώ, δεν είμαι μηχανικός επικοινωνιών. η βαθύτερη αξιολόγηση κινδύνου θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες μετά τη νέα μελέτη που σας προανέφερα. Βεβαίως η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη τώρα με σημαντικά κονδύλια την έρευνα για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αυτό το κάνουμε εδώ και χρόνια και με το προηγούμενο και στο μέλλον. Με το προηγούμενο και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Αφού ακούσαμε την Επιτροπή και τα μέλη που μίλησαν και από το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές και τους πράσινους που όλοι ζήτησαν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά προτείνω να μην ανοιχτεί αναφορά, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας στείλει όταν έχουν τις πληροφορίες, να μας ενημερώνει τέλος πάντων την έκθεση του ICNIRP e που θα δημοσιευθεί σε λίγο καιρό, καθώς και τις μελέτες που κάνει η Επιτροπή για τον αντίκτυπο του 5G ό,τι κάνει τέλο πάντων το ICNRP και να συνεχίσει να υποστηρίζει με κονδύλια της Επιτροπής ε, την έρευνα για τις νέες αυτές τεχνολογίες. Η Επιτροπή είπε ότι έκανε ε, ε, ε, έχει χρηματοδοτήσει μελέτες για την ναι, αυτή την τεχνολογία. Ζητώ από την Επιτροπή να μας στείλει λοιπόν όχι μόνο την ενημερωμένη έκθεση του ICNIRP, e όχι μόνο τις μελέτες αντικτύπου που κάνουν για τον πληθυσμό, συνολικά τον πληθυσμό, όχι μόνο τις ευάλωτες ομάδες, για τα 5G και τα προγράμματα που υλοποιεί για το, τα 5G. Οι σοσιαλιστές επίσης μου ζήτησαν να στείλουμε και την αναφορά στην Επιτροπή ΕΜΒΗ που είναι πιο αρμόδια στο θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Ωραία, ευχαριστώ όλους. Επόμενο σημείο, 21. Αναφορά 477-2019 του Γκουστάβου Αλντόλφο Σεράνο Ιδάλγκο, Ισπανού πολίτη, εξ ονόματος ε, του, της Ένωσης National Nemesis Project για την ε, ρύθμιση της χρήσης της κανάβεως. Καλωσορίζω τον αναφέροντα. Έχετε πέντε λεπτά για να παρουσιάσετε την αναφορά σας, μετά η Επιτροπή, μετά τα μέλη και αν θέλετε κύριε Κατόπιν, ε, κύριε Ιδάλγκο, θα έχετε και δύο λεπτά στο τέλος. Καλωσορίσατε και σας δίνω το λόγο. Τώρα μπορώ, ε. Πολύ ωραία. Εκπροσωπώ την ε, Ένωση Σχεδίου Νέμεσης ε, για την ε, ρύθμιση της νόμης χρήσης Κανάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ισπανία, στη Βουλή, ζητάμε να υπάρχει μια νομοθετική πρωτοβουλία για να ρυθμίσουμε την ασφάλεια, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών στη Μικτή Επιτροπή για τη Μελέτη του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ισπανία υπάρχει ένας ε, νόμος ε, που προκύπτει από το 67, που προκύπτει από την ε, έκθεση των Ηνωμένων Εθνών το 61 και ρυθμίζει τη χρήση ναρκωτικών και ψυχότροπων νησιών. Υπάρχουν θέματα για ασθένειες χωρίς να υπάρχει φαρμακευτική απάντηση η παράνομη χρήση και η διαφορά με την ελεγχόμενη χρήση και η παραγωγή φυσικής κανάβεως για ιατρική χρήση και όλα αυτά για τη δημιουργία του Ισπανικού οργανισμού που ρυθμίζει την προστασία και την ε, υπεράσπιση των ατόμων για τα θεμελιώδη δικαιώματα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα αυτά θα προωθήσει την ε, προοπτική της Ισπανίας και θα βοηθήσει στην προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ε, προσπαθώντας να έχουμε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών. Θέλουμε να προστατεύουμε και να ρυθμίζουμε τη χρήση κάναμες. Συγγνώμη, πώς μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί έτσι θα διευκολύνουμε και τη διαρμηνία. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο σκοπός της Ισπανικής Υπηρεσίας, βέσω τη οποία ρυθμίζεται η προστασία ε, και η υπεράσπιση των θεμελιών δικαιωμάτων των πολιτών και τις σχέσεις τους με τις ε, δημόσιες διοικήσεις, έχει ως στόχο την επιστημονική υποστήριξη και την έρευνα για τον αντίκτυπο των προϊόντων ε, που προέρχονται από την κάναβη. Θα υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα βασίζονται στην ιατρική κατάρτιση και στην κατάλληλη ενημέρωση ε, και θα προωθήσει την φαρμακευτική κάναβη ε, και θα ε, δούμε και τι έχει γίνει γιατί υπήρξαν εφάλματα τα οποία σχετίζονταν από τις ελλειπείς ιατρικές γνώσεις και πληροφορίες για τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση σε συγκεκριμένα θεραπεία και πάλι τα νέα στοιχεία θα τα λάβουμε ε, από την ε, παράνομη κατανάλωση που ε, γίνεται εδώ και χρόνια και την παρακολουθούμε εδώ και χρόνια και βλέπουμε τι γίνεται με τη δραστική ουσία που ανταποκρίνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη παθολογία. Έτσι θα έχουμε τις διαφορές μεταξύ ψυχαγωγικής και θεραπευτικής χρήσης. Επίσης θα δούμε και τη σημασία και την ανάγκη να υπάρξει κατάλληλη χρήση των προϊόντων που βασίζονται στην κάναβη και θα πρέπει να δώσουμε μάχη για μια νοτροπία η οποία υπάρχει εδώ και 70 χρόνια. Υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν να χρησιμοποιούνται για ε, χρήση και κοιτάμε να δούμε και τι γίνεται και ο οργανισμός που θέλουμε να δημιουργήσουμε θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο να βρούμε μέτρα όταν θα πρέπει να δούμε ε, εάν έχουν ε, παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον αντίκτυπο της κάναβης και επιμένως ε, δεν θα πρέπει να ευνοήσουμε σε καμία περίπτωση τα δίκτυα εμπορίου ναρκωτικών και ε, να βοηθήσουμε τη χρήση. Θα πρέπει οι παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να γίνουν νόμισμες δραστηριότητες και θα ε, περάσουν στους ε, επίσημους μηχανισμούς και θα, ε, δεν θα είναι οι έμποροι αυτοί που θα ελέγχουν τα πράγματα, αλλά θα είναι οι ιατροί και εξειδικευμένο προσωπικό. Θα γίνεται λοιπόν χρήση με ελεγχόμενο τρόπο. Θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη από τους ανηλίκους και τους νέους που βλέπουν στην κατανάλωση κάναβες ότι είναι ε, μέρος της ε, κοινωνικής τους ψυχαγωγίας. Οι ευάλωτοι είναι αυτοί οι νέοι που θεωρούν ότι η χρήση κάναβες είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουν την προσοχή των άλλων, προσελκύσουν προσοχή άλλων ανθρώπων ε, και αλλιώς δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν απαντήσεις που, και αποφάσεις οι οποίες ε, είναι από πιέσει του κοινωνικού του περίγυρου. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προτεραιότητα για οποιοδήποτε εθνικό οργανισμό και ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίο ε, ε, θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι βασικές αξίες που μας κάνει πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βλέπουμε τους, τους χρήστες στα εγκεκριμένα κέντρα και με τις άλλες ναρκωτικές ουσίες. Και ορισμένες φορές έχουμε κατανάλωση και άλλων ουσιών, χρήση και άλλων ουσιών και πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι χρήστες που πηγαίνουν σε κέντρα αποτοξίνωσης είναι άτομα τα οποία έχει στείλει η δικαστική εξουσία ε, για να μην ε, βρεθούν στη φυλακή και είναι η εναλλακτική λύση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στα κέντρα αποτοξίνωσης και πραγματικά υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την περίπτωση. Η Ισπανική υπηρεσία που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ως στόχο να παρουσιάσει βάση ε, πρωτοβουλειών των πολιτών τα άρθρα τα οποία θα πρέπει να τελειώσετε κάποια στιγμή διότι ε, έχετε ε, υπερβεί το χρόνο. Αν μπορείτε να ολοκληρώσετε λοιπόν. Μετά από όλα λοιπόν όσα σας διάβασα η ρύθμιση της χρήσης ε, και κατανάλωσης κάναβης ε, και η διαδικασία της ε, ανανέωσης του νόμου του 67 Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τον τρόπο να συσταθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που θα έχει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ίδιο δίκτυο που θα ρυθμίζει τη χρήση κάναβης. Ευχαριστώ. por parte Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεράνο Ιδάλγο για την αναφορά του στο θέμα αυτό. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε πλήρη επίγνωση του ζητήματος και της βαρύτητας της κάναβης και της χρήσης ε, ε, στο φαρμακευτικό τομέα θα δώσω το λόγο στην άδελφο Άγνες Ματιού στη συνέχεια. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο αφορά το εξή. Η Διεθνή Σύμβαση για τα Φάρμακα ε, εμπέπτει στον ε, νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 8 που αφορά τα σκευάσματα τα οποία εμπέπτουν στον έλεγχο της Σύμβασης ε, των Ηνωμένων Εθνών του 2017 και η κάναβης ε, εμπίπτει σε αυτή την ε, νομοθεσία. Ε, θεωρείται, ε, ελέγχεται λοιπόν η κάναβης από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Ε, είναι νόμιμη χρήση της για επιστημονικούς σκοπούς και για φαρμακευτική χρήση, αλλιώς είναι παράνομη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς σκοπούς. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η προσεγγίση των χωρών μελών ε, και όσον αφορά τον έλεγχο της πολιτικής των ε, ναρκωτικών ε, διαφέρουν και στο βαθμό αυτό οι προσεγγίσεις των χωρών μελών για την κάναβη ευθυγραμμίζονται με την σύμβαση. Ε, καμιά από τις χώρες αυτές δεν έχει νομιμοποιήσει την κάναβη για προσωπική χρήση, για μη φαρμακευτική χρήση και θα ήθελα να θέσω στην Επιτροπή Αναφορών το εξή ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αξιολογεί τη στρατηγική για τα ναρκωτικά. Έχουμε την ε, στρατηγική από το 12 έως το 20. Εάν ενδιαφέρεστε για το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω ότι, είναι πρόσδεκτη η εισφορά του αναφέροντα για το θέμα αυτό σε οποιαδήποτε από τις ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε και εμείς, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποια πρόταση και να κάνει θα πρέπει να είναι στην ίδια γραμμή με την ε, Συμβέση των Ηνωμένων Εθνών. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο Ματιό για να εξηγήσει το ζήτημα της Κάναντης και τη φαρμακευτική χρήση. Θα ήθελα να αυτό στη φαρμακευτική χρήση της κάναβης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ε, στέρεο ε, ε, νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την φαρμακευτική χρήση της κάναβης. Και εμπίπτει η χρήση κάναβη σε αυτό το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν βλέπουμε το λόγο να υπάρξουν εδώ εξαιρέσεις. Αυτή στιγμή παράγεται ένα νέο σκεύασμα, θα πρέπει η εταιρεία να παράσχει τα δεδομένα που να αποδεικνύουν την ασφάλεια του ε, σκευάσματος και την αποτελεσματικότητά του για την πρόληψη κάποιων ασθενειών. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ε, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούν να αποδείξουν ακριβώς την ποιότητα και την ασφάλεια αυτών των σκευασμάτων. Ε, όσον αφορά τη κάναβη, ε, χρησιμοποιείται για την επιληψία και, τους, ε, και διάφορες μυοπάθειες, μυϊκούς σπασμούς και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η νομοθεσία επιτρέπει και καταδεικνύει ότι είναι δυνατόν τα σκευάσματα αυτά να λανσαριστούν στην αγορά υπό τη φαρμακευτική τους ιδιότητα. Η Επιτροπή Αναφορών ε, τονίζει το ρόλο της ε, αίμα, η οποία ε, αξιολογεί την ποιότητα των σκευασμάτων. Ένα από αυτά τα σκευάσματα έχει εγκριθεί, έχει αξιολογηθεί από την ΕΜΑ και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίση να διευκρινίσω ότι η ταξινόμηση των προϊόντων αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των χωρών μελών, εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα να αξιολογήσουν κατά πόσο η κάναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φαρμακευτική χρήση και επίσης οι χώρες μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι η νομοθεσία περί φαρμάκων είναι δεδειγμένη ή όχι, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια παρέκκληση από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και μια χώρα μπορεί να επιτρέψει τη χρήση προϊόντων ε, αλλά υπό τον αυστηρό έλεγχο εμπειρογνώμων ε, του κλάδου υγείας με την εξήγηση αυτή μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε ότι η νομοθεσία για τα φάρμακα είναι δεδειγμένη όταν έχουμε ένα προϊόν το οποίο βασίζεται στην κάναβη προκειμένου να, δοθεί, να χορηγηθεί έγκριση για τη χρήση του σε ασθενείς ή κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν παρεκκλήσεις από χώρες μέλη ε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η κατα ποσο μπορουν να εφαρμοστουν παρικλησεις απο χωρες κάναβης. Ε, τέλος, αναφέρθηκε η δυνατότητα για τις χώρες μέλη να υπάρξει εκπαίδευση και επαρχή βοήθειας προς τους νέους ανθρώπους και θα ήθελα να ευκρινίσω ότι η οργάνωση του συστήματος ε, περίθελψης ε, και υγείας εμπίπτει στις χώρες μέλη, οι οποίες μπορούν αυτές να αποφασίσουν πώς οργανώνουν την υγεία στη δική τους επικράτεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαλίβα. πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε για την φαρμακευτική χρήση της κάναβης τη δυνατότητα πρόσβασης στην φαρμακευτική αγορά στα κράτη-μέλη. Θυμίζω ωστόσο και ένα ψήφισμα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στι 13 Φεβρουαρίου του 2019 που ζητούσε από όλα τα κράτη-μέλη να παρεξετάσουν τη σχετική νομοθεσία για τη χρήση ε, φαρμάκων βάση που βασίζονται στην κάναβη εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να, χρησιμο... να, να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα με άλλα παραδοσιακά φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την διαδικασία αυτή αναμένοντας άλλες πληροφορίες από την Επιτροπή και να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης, ώστε οι ασθενείς ανά την Ευρώπη να μπορούν να κερδίσουν από τις θετικές συνέπειες ε, που φάρμακα που βασίζονται στην κάναβη μπορεί να φέρουν στη μείωση του πόνου στους ασθενείς στην Ένωση. Βίντσεν. Και εγώ ξεκινώ θυμίζοντας το ψήφισμα που εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο στις αρχές ε, του προηγούμενου έτους για την χρήση της ε, κανάβεως για φαρμακευτικούς λόγους που ζήτησε από τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν την ε, νομοθεσία τους σχετικά εφόσον επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα φάρμακα. Εμείς όπως εμείς κάναμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, είδαμε και ότι η Επιτροπή έχει τη δική της προσέγγιση στον τομέα αυτό. Βέβαια το θέμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση στην Ένωση για το θέμα αυτό. Ως ΕΛΚ θα προτιμούσα λοιπόν να κλείσει η αναφορά. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για τον αναφέροντα, για να κλείσει. Ευχαριστώ. Το 2015, ο ΙΕ, το Μάρτιο του 2015, ο ΙΕ εξέδωσε μία έκθεση που έλεγε ότι απέτυχε το σύστημα καταπολέμησης των ναρκωτικών. Αυτό πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, μία, με ένα ψήφισμα μη δεσμευτικό που έλεγε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να δημιουργήσουν εθνικές επιτροπές ούτως ώστε να μπορούν ομάδες ή δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουν μέσω των κρατών μελών τους 5-6 υπηρεσίες πάντων σε κάθε κράτος να μπορούν να συνεδριάσουν για να υιοθετήσουν δεσμευτικές αποφάσεις. Τα κράτη αποφασίζουν, αλλά ενωμένα, μαζί, προς μία κατεύθυνση, τη ρύθμιση, να υπάρξουν αποτελέσματα για τα άτομα που πάσχουν και που χρειάζονται μία φαρμακευτική αντιμετώπιση με βάση φάρμακα που στηρίζονται σε κάναβη. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού ακούσαμε τον αναφέροντα, την Επιτροπή και τους βουλευτές, το λέω προς τον αναφέροντα ότι εμείς προσπαθούμε να αποφασίσουμε πάντα με βάση και το τι φρονούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ε, το ΕΛΚ ζήτησε να κλείσει, οι σοσιαλιστές ζήτησε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Η πρόταση της Προέδρου βάσει και αυτόν που είπε επί το οποίο ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που έχουν την αρμοδιότητα να νομοθετούν για το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να νομοθετεί για την θεραπευτική κάναδη και ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει θέση με ένα ψήφισμα, προφανώς δεν έχει αρμοδιότητα, είπαμε η αρμοδιότητα των κρατών μελών, στις 13 Φεβρουαρίου του 19 ωστόσο το Κοινοβούλιο πρότεινε πέρασε ένα ψήφισμα για τη χρήση της κανάβεως για θεραπευτικούς λόγους. Η πρόταση της Προεδρίας είναι να κλείσει η αναφορά λόγω έλλειψης αναφοράς. Η Επιτροπή είπε ποια είναι η αρμοδιότητα των κρατών μελών και άφησε, κατέστησε σαφές προ τον αναφέροντα, καθιστούμε σαφέ στον αναφέροντα ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί με το θέμα με ένα ψήφισμα. Παραπέρα δεν μπορούμε να πάμε. Δεν έχουμε άλλες αρμοδιότητες. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και ευχαριστώ την Επιτροπή για την απάντησή της. Περνάμε τώρα στο σημείο 22. Τέσσερις αναφορές έχουμε εδώ. 299-2018, 1124-2015, 18-2019 και 435 του 2019 από Ισπανούς, Βρετανούς και Ιταλούς πολίτες για τη διάκριση μεταξύ φίλων σε θέματα ε, φύλου για μείωση του ΦΠΑ στο 0% για προϊόντα γυναικείας προσωπική υγιεινή ε, και κατάργηση το 22% ΦΠΑ για πάνες και άλλα προϊόντα και ε, μείωση του φόρου για σχετικά αντίστοιχα προϊόντα. Επειδή δεν υπάρχει κάποιος από τους αναφέροντε εδώ στην αίθουσα, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Άλβαρο Ολιβέηρα από τη Γενική Διεύθυνση Just. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με την άδειά σας θα μιλήσω αγγλικά. Δεν υπάρχουν εδώ παρουσία αναφερόντων και θα ήθελα να πω ότι ζητούν την κατάργηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του λεγόμενου ροζ φόρου, τουλάχιστον στην πρώτη αναφορά ε, για την οποία ε, παρουσιάζω τη θέση μας, λένε ότι υπάρχει μια επιπλέον επιβάρηση για τις γυναίκες για κάποια προϊόντα ή κάποιες υπηρεσίες τα οποία διατίθεται στο εμπόριο για γυναίκες ειδικά ε, και είναι όμως πανομοιότυπα στην ουσία με προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο για άντρε. Εγώ προσπαθώ να σπάσω λίγο τον, και να, τον πάγο και να τα θέσω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο και θα αναφερθώ στην ισότητα μεταξύ ανδρών και ε, γυναικών και οι συνάδελφοι από τη Γενική Διάθεση Ταξούντ θα αναφερθούν στο πιο σημαντικό θέμα του φόρου τη Θεμενή αξίας και τη σχετική οδηγία. Να υπενθυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει οδηγία του 2004 κάθοτος 113, η οποία απαγορεύει την άμεση και έμεση διάκριση σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και προμήθειά τους. Για να πάρω το παράδειγμα της πρώτης αναφοράς, το γεγονός ότι ένα προϊόν υποτίθεται ότι είναι για άνδρες, για παράδειγμα ένα ξηραφάκι σε μπλε χρώμα, το γεγονό ότι αυτό το ξηραφάκι θα μπορούσε να είναι φτηνότερο από το αντίστοιχο ξηραφάκι ε, σε ροζ εκδοχή, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο για γυναίκε, δεν σημαίνει απαραίτητο ε, ότι πρόκειται για διάκριση βάση φύλου και ε, επομένως θα ισχύει η οδηγία. Αυτό ισχύει μόνο εάν το ίδιο προϊόν προτείνεται σε διαφορετική τιμή για άνδρες και γυναίκες. Αλλά όπως σας είπα, αυτό ήταν ε, απλώ η εισαγωγή και από εκεί και πέρα με την άδειά σα θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου μα από τη Γενική Διευθυνσία Ταξούντ. Ναι, ο κύριος Μικελέτο. First of all, I'm sorry. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, ε, ζητώ συγγνώμη που μιλάμε για τις διακρίσεις. Εγώ είμαι άντρα και μιλάμε για διακρίσεις κατά των γυναικών. Δεν έχουμε όμως γυναίκα συνάδελφο. Το θέμα είναι δική μου αρμοδιότητα. Δυστυχώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχει οδηγία ΦΠΑ 2006-112, η οποία στο άρθρο 98 και πάλι και στο παράρτημα 3 αναφέρει ένα κατάλογο προϊόντων για τα οποία υπάρχει δυνατότητα ε, για μειωμένο ΦΠΑ. Τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται εκεί είναι προϊόντα για τα οποία τα κράτη-μέλη επιτρέπεται ε, να χρησιμοποιήσουν αυτό το ενδεχόμενο. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν ε, εφαρμόζουν μειωμένο ΦΠΑ και κάποια άλλα δεν εφαρμόζουν μειωμένο ΦΠΑ και δεν εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει μια κάποια διαφοροποίηση, αλλά αυτό επιτρέπεται από την οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιανουαρίου του 2018 πρότεινε να επανεξετάσουμε το τομέα του μειωμένου ΦΠΑ. Και στο άρθρο 98, την αναθεώρηση του άρθρου 98, λέγεται σαφώς ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένο συντελιστά στη ΦΠΑ ε, κατώτερο από το 5%, δηλαδή ακόμα και το 0 που ζητούσε κάποιος σε κάποια αναφορά. Πρόκειται όμως για μια πρόταση, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συζήτηση στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, ε, επιτρέπεται όμως τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε κάποια προϊόντα και ε, προϊόντα ε, προσωπικής υγιεινής, αν το επιθυμούν. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Να πω μόνο ότι χαίρο που πέβαλαν δύο Ιταλοί την ε, αναφορά αυτή. Είναι μία, δύο Ιταλίδες μάλλον την αναφορά αυτή. Είναι ε, αναφορές που θέτουν ένα ζήτημα πολύ δίκαιο πολλές χώρες της Ένωσης εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα μείωσης του συντελεστή, άλλοι δεν το κάνουν. Η δική μου ευτυχώς το έκανε στο τελευταίο προπολογισμό που μείωσε το συντελεστή στο 5%. Δύο πράγματα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει μία ξεκάθαρη ένδειξη. Το καταλαβαίνω αυτό. Θα ήταν καλό ωστόσο, απευθύνομαι στους δύο κυρίους, αλλά αφορά όλου. Θα ήταν σκόπιμο να δώσει κάποια μηνύματα η Επιτροπή καλώντα τα κράτη, προτείνοντα η καλή αυτή πρακτική να γίνει πρακτική όλων. Δεύτερον, πέραν του θέματος του carbon tax, του, ε, του, του, του, του φόρου ε, φόρου για τα ταμπών, χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα τα ζητήματα των προϊόντων γυναικείας υγιεινής. Το να περιορίζουμε λοιπόν ε, το θέμα μόνο σε ένα συγκεκριμένο προϊόν που σε κάποιες χώρες είναι ε, σε προϊόντα που μπορεί σε κάποιες ε, ε, κατηγορίες ε, οικογενειών να είναι προβληματικά οικονομικά, θα έλεγα ότι σε πολλές οι πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι όντως η οικογένεια, η μητρότητα είναι σημαντικά και το θέμα των πανών είναι ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα που θα έπρεπε να εξετάσουμε. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να φροντίσουν ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν το ζήτημα και να ε, το δουν με έναν πιο ανοιχτό τρόπο. Ευχαριστούμε. Κύριος Βίντσε, ευχαριστώ την συνάδελφο για τις εξηγήσεις που δίνει. Πιστεύω ότι καλύτερα είναι να το κάνει η ίδια. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω και εμείς ως Επιτροπή πρέπει να στραφούμε. να κλείσουμε, να την αφήσουμε ανοιχτή δεν ξέρω, αλλά η τάση μου είναι μάλλον να μην είναι ανοιχτή η αναφορά. Εμείς πάντως είμαστε ανοιχτοί, ας δούμε και τι θα έρθει από την Επιτροπή. Βέβαια, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να αναλάβουν δράση κατά βάση. Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις της Πατρίτσια Τόια. Ως σοσιαλιστές ζητούμε να μην ανοιχτεί η αναφορά. Και εμείς υποστηρίζουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα ήθελα σαφέστες απαντήσεις από την Επιτροπή τι κατηγορίες προϊόντων μπορεί να προτείνει να χρησιμοποιηθούν για να επεκταθεί το παράδειγμα της οδηγίας. Έχετε κάνει κάποιες μελέτες, προτάσεις για το θέμα αυτό. Η κυρία Κώσα. Ο κύριος Κώσα. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές και θέλω να τονίσω ότι είναι προφανές ότι όσοι γνωρίζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζουν ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Είναι σκόπιμο επίσης να καταλάβουμε ότι τα προϊόντα αυτά είναι αναγκαία για τις γυναίκες. Πρέπει ωστόσο να αποφύγουμε την παγίδα να βάλουμε κάποιες κατηγορίες μπροστά από άλλες. Για παράδειγμα, αν δούμε τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία. Πάντα υπάρχουν ομάδες που ζητούν μέτρα για την προστασία της κατάστασής τους. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν προσεκτικά εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε έχοντας ακούσει την Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής μας. Κρατάμε ανοιχτή την αναφορά. Ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο για το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά ιδίω αυτά τα προϊόντα. Σημείο 23. Γνωμοδότηση για τον έλεγχο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του 2017 και 2018. Σοσιαλιστής είναι ο εισηγητής προς γνωμοδότηση, το Ρουίς Ντεβέζ, ο οποίος έχει καθυστερήσει γιατί έχει κακοκαιρία στην ε, Ισπανία όπως ξέρετε. Δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Είτε να μας μιλήσει ο κύριος Σαλίβα αντί για τον εισηγητή ή το αναβάλουμε το απόγευμα. Μην ξεχνάτε όμως ότι το απόγευμα έχουμε πολλές ε, αναφορές. Τι έχετε να πείτε κύριε Σαλίβα. εκ μέρους του Ντομινίκ Ρουίς Τεβέσα. Θα διαβάσω τις δηλώσεις του. Αυτή η γνωμοδότηση έχει σαν στόχο να υποβάλει κάποιες ιδέες όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας το 17 και το 18. Η γνωμοδότηση αυτή αξιολογεί τα δικαιώματα των ε, πολιτών ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ένας, ένας ε, πολύ ξεκάθαρος μηχανισμός όσον αφορά την ε, παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση για την εφαρμογή του κράτους δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Υπάρχει αύξηση του αριθμού αναφορών από πολίτες για περιπτώσεις παραβίασης ε, του κράτους δικαίου, αύξηση καταγγελιών 3.850 το 2018. Η μεγαλή ο μεγαλύτερος αριθμός των καταγγελιών αυτών έχουν αποσταλεί στην ε, Επιτροπή. Ε, στην έκθεση του 18 υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και επισημαίνεται ότι στις περισσότερες αυτές αναφορές η Επιτροπή δεν έχει κινήσει μια διαδικασία εξέταση, έχει λάβει άλλα μέτρα όσον αφορά το περιβάλλον, τη μετανάστευση, την ελεύθερη διακίνηση και την ε, φορολόγηση. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα. Από την έννοια αυτή ζητούμε από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς μπορεί να λύσει το χάσμα αυτό μεταξύ των ε, παραπώνων και καταγγελιών που έχει λάβει και της έλλειψη λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι τον 28 ε, Ιανουαρίου στις 3 ώρα το μεσημέρι. Perfecto. Ωραία, λοιπόν. Ο κύριος Σώσα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Ντεβέσα για την εργασία του. Ε, λυπούμε που δεν ε, βρίσκεται εδώ σήμερα, αλλά ελπίζω ότι αυτά που θα του θα πω τώρα, εξ του ΕΛΚ, θα του διαβιβαστούν. Έχω κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν αυτή την γνωμοδότηση. Είναι αναγκαίο να μιλείς, να γίνει συζήτηση για τις καταγγελίες των Ευρωπαίων πολιτών και να προβούμε στην εξέβρεση λύσεων. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την ε, το χώρο για την ε, χρήση πολιτικών ε, δηλώσεων. Θα πρέπει να παραμείνουμε αντικειμενικοί. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αφιερθεί μια ολόκληρη παράγραφο στο ζήτημα του κράτους δικαίου, έστω και αν ε, η θεμελιώδης αρμιοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών είναι να διαχειρίζεται τις αναφορές. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να περιγράψουμε την κατάσταση βεβαίως υπόρους επικορικότητας. Τα... Η αναφορά αυτή μπορεί να επιληθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε μη εθνικό επίπεδο. Αναμένω την συνεργασία σας και ελπίζω ότι θα συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση δική μας άποψη και θα διαβιβαστεί στην Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Γι' αυτό θα κλείσουμε εδώ. El ponente Ruiz de Ο κύριος δεν ε, μπόρεσε να παρέμβει, μίλησε ο κύριος ε, Σαλίβα, αλλά τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Βασικά αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημώνω εδώ για το σχέδιο γνωμοδότησης είναι ότι συνενώνει το συμβασμό της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία της εφαρμογής του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης τη Βούλη συναγγηθεί η διαφάνεια για πολλές αναφορές που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δράσεις παρακολούθησης. Ως... Ε, επίσης υπάρχει μια άλλη πτυχή την οποία θα ήθελα να επισημάνω στους συγητής που αφορά το δικό μου συμβιβασμό, ε, ούτως ώστε η αυτή να επισημάει, να τονίσει την ανάγκη προάσπισης του κράτους δικαίου, ρουλοφλό και των εγγύσεων ε, εφαρμογής της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό θα μοιάζε μη αναγκαίο, περιττό σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς οι απειλές οι οποίες ε, αφορούν την μη εκπλήρωση του κράτους δικαίου σε πολλές χώρες μέλη, καθιστά αναγκαία και επιτακτική την ανάγκη να υπογραμμίσουμε την απέτηση εκπλήρωσης των εγγύσεων υπέρ των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η μη εκπλήρωση της εφαρμογής ε, του δικαίου αυτού όχι μόνο έχει επιπτώσει στον, στην εσωτερική αγορά, αλλά επηρεάζει σημαντικά την αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας ε, το, τις τάσεις εθνικισμού και λαϊκισμού οι οποίοι ε, ε, προσπαθούν να υπονομεύσουν το κράτος ε, δικαίου και τις απαιτήσει αυτές που απορρέουν από αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω την γνωμοδότησή μου και να επισημάνω τα μέσα που έχουμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες μέσω εξεταστικών επιτροπών στο επίπεδο των χωρών μελών που να συμπεριλαμβάνουν τις ανησυχίες των πολιτών. Αξιολογούμε θετικά το έργο του εισηγητού, αλλά θέλαμε, θέλουμε μια κίνηση για την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου ως μοναδικού τρόπου να ε, προωθηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσπίζει τα δικαιώματα των πολιτών ε, και προώθησης των δημοκρατικών αξιών του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα θα πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια εποπτείας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη και πάλι για την καθυστέρησή Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας ε, για την παρουσίαση αυτής της γνωμοδότησης. Η εφαρμογή των αρχών αυτών αποτελεί προτεραιότητα και πιστεύω ότι φυσικά πρέπει να προστατεύουμε αυτές τις αρχές. Ε, βέβαια πάντα μπορεί να βελτιωθεί η εποπτεία θα ήθελα να προτρέψω τους πολίτες να ε, υποβάλουν αναφορές, ε, διότι μόνο έτσι μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή μας. Ε, αναφορές θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Ε, γνωρίζω πολλούς από τους αναφέροντες, ε, τους έχω γνωρίσει εδώ και όταν έχουμε την απαραίτητη αρμοδιότητα αναζητούμε ένα τρόπο να βρούμε μια λύση ή τουλάχιστον να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συντάκτη της γνωμοδότησης και να ευχαριστήσω και τους ε, σκιώδεις συντάκτες. Αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα δεν γίνονται πάντα αντιληπτά όπως θα έπρεπε και δεν ε, δημοσιοποιούνται και όπως θα έπρεπε. Η διαφάνεια είναι όρος που είναι της μόδας, αλλά οι πολίτες ε, θα πρέπει να γνωρίζουν και τι γίνεται στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να λογοδοτούμε στους πολίτες μας και ο εισηγητής ε, αναφέρεται στη διαφάνεια και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε διότι οι πολίτες μας το αξίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Ρενέ Σλότιες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σχολιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, ξέρω ότι θα υποβληθούν και τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο γνωμοδότησης, διότι επισημαίνει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος ε, στην έκθεση του 2018 για τη διαφάνεια. Επομένως, δίνουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες ε, και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι κάνουμε εμείς και όχι μόνο για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Άκουσα κάποια σχόλια, επομένως απλώς θα σχολιάσω ακροθυγώς κάποια εξ αυτών αν μου επιτρέπετε. Για μα ε, φυσικά η αποτελεσματική εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εφαρμόζεται σωστά για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Κομισιόν και είναι και πολύ σημαντικό όσον αφορά το κράτο δικαίου και φαίνεται άλλωστε και από την αποφασιστική και γρήγορη δράση που αναλάβαμε για κάποιε απειλέ για την ανεξαρτησία των δικαστηρίων σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι δημόσιο βεβαίω. δεν θα πω κάτι περαιτέρω για τους αναφέροντες. Ε, ναι, φυσικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, θέλουμε να δούμε πολύ περισσότερες πληροφορίες ε, επ' αυτού στις ετήσιες εκθέσεις μας ε, και θα εξετάσουμε από κοινού με την Επιτροπή και τη Γραμματεία πώς μπορούμε στην πράξη να κάνουμε κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις για την ετήσια έκθεση, πώς θα μπορέσουμε να δίνουμε περισσότερα στοιχεία για τις αναφορές που επεξεργαζόμαστε Επίσης, ε, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πλέον αρμόδια για να δει ε, διαρθρωτικές παραβιάσεις ε, που καλύπτουν μεγάλο αριθμό πολιτών. Δεν έχουμε όμως τους πόρους να εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γι' αυτό ακριβώ, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο της γνωμοδότησης, σε πολλές περιπτώσεις παραπέμπουμε τους αναφέροντες σε άλλα όργανα, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο επίλυσης διαφορών ή και το σόλβιτο για να επιλύσουν το πρόβλημα όπου μπορούν, διότι πρώτον δεν υπάρχουν κατάλληλοι πόροι και δεύτερον είναι πολύ καλό και για τους πολίτες, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη η επίλυση του προβλήματος η ε, διαδικασία επί παραβάση δεν έχει στόχο να προσφέρει λύση ενός προβλήματος, αλλά ε, να ε, τιμωρεί στα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να δώσουμε αποζημιώσεις στους πολίτες για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, για παράδειγμα, ή να υπάρχουν συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις. Οι διαδικασίες επί παραβάση, όπως έχουν δημιουργηθεί, είναι χρονοβόρες και αυτό φυσικά πρέπει να το έχουμε και κατά νου είναι απλώς ε, θέμα επικουρικότητας. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα επιλύονται πολύ καλύτερα πιο κοντά στον πολίτη και πιστεύουμε ότι είναι και προς το συμφέρον του. Βεβαίω, ε, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ε, εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυση διαφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να διεκπεραιώνει αυτέ τι καταγγελίε. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη διαφάνεια των αναφορών. Ευχαριστώ και το συντάκτη και τους κοιόδες συντάκτες και την Κομισιόν για την παρέμβασή της. Να σας πω απλώς ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 28 Ιανουαρίου του 2020 στις 3 η ώρα. Κλείνει λοιπόν η συνεδρίαση για σήμερα το πρωί και σας περιμένουμε στις 2.30 που θα συνεχιστεί η συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.